μονάδες. Ο κύριος Λένε, ο εισηγητής, έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην έκθεση αυτή πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο εδώ και πολλά χρόνια απασχολεί το Κοινοβούλιο και τώρα γίνεται ένα περαιτέρω βήμα προς την επιτυχία αυτού του προγράμματος. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρομονάδες και εδώ εννοούμε τις πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις με πολύ λίγους απασχολουμένους, με μικρό κύκλο εργασιών και κυρίω είναι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και έχουμε κατά νου το φούρνο, το μπακάλι, τέτοιου είδου ε, επιχειρήσει που θέλουμε να απελευθερώσουμε από μεγάλο διοικητικό φόρτο. Το Κοινοβούλιο πολλέ φορέ προσπάθησε σε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, επανεξετάζοντα την 4η και την 7η οδηγία, να ε, εφαρμόσει κάτι για τι μικρομονάδε. Και σε αυτό το πλαίσιο ε, υπάρχει η έκθεση του συναδέλφου Βάντερμπουργκ στο τέλο του 2008, αλλά δεν καταλήξαμε τελικά με το Συμβούλιο να το θέσουμε σε λειτουργία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 2008 υπέβαινε ένα ψήφισμα όπου σχεδόν ομόφωνα πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς αυτή τη δυνατότητα της απελευθέρωσης των ε, μικρομονάδων ε, να την εφαρμόσουμε. Στο μεταξύ, ακριβώ αυτό γίνεται. Υπέβαλε μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνοντα ακριβώ αυτό το οποίο ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε την ομάδα Stoiber για να ασχοληθεί με τα προβλήματα αυτά και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και απεφάνθη ότι είναι αποφασιστικό εργαλείο για να ε, απαλλαγούν από την ε, γραφειοκρατία οι μικρομονάδες και μιλάμε για εξοικονόμηση 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν ε, η άρση της επιβάρυνσης για τις μικρομονάδες. Είναι η ναυαρχίδα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από τις γραφειοκρατικές ε, διατάξεις. Αυτή η οδηγία για την οποία μιλάμε είναι μια οδηγία του 1978. Είναι μια επιτροπή η οποία βασίστηκε στις μεγάλες και τις μεγάλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποτέ αυτή η οδηγία δεν αφορούσε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις μικρομονάδες. Μέσω αυτής της οδηγίας ε, προτείνεται η σύνταξη ισολογισμών ε, και αιτησίων λογαριασμών που ε, είναι που έχουν ε, δημιουργηθεί για τις μεγάλες επιχειρήσεις και σίγουρα όχι για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μια τόσο μικρή επιχείρηση, αν χρειάζεται ε, ε, πιστώσεις, θα έπρεπε να υποβάλει όλα αυτά τα στοιχεία του ισολογισμού, ενώ οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα και με τις έρευνες της Επιτροπής, δεν γνωρίζουν καν το πώς καταρτίζεται ο ισολογισμός. Επομένως, δεν έχει καμία αξία για τις μικρομονάδες τη διάταξη. Αυτό που έχει σημασία για τις μικρομονάδες ε, είναι το cash flow και η ρευστότητα. Αυτό μας ενδιαφέρει για τις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις ε, μικρομονάδες. Μας ενδιαφέρει να δούμε αν υπάρχει ρευστότητα στις επιχειρήσεις αυτές για να μπορέσει να καθοριστεί το θέμα της λήψης πιστώσεων από τις επιχειρήσεις αυτές. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν ε, έχουν επιπτώσει στις διαμεθοριακές συναλλαγές. Επομένως δεν έχουν επίπτωση σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτές οι επιχειρήσεις ε, ε, δραστηριοποιούνται σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, συνήθως μέσα στο ίδιο το κράτος μέλος. Αυτές οι διατάξεις αφορούν περισσότερο διασυνοριακά τις εταιρείε που έχουν επίπτωση στην ενιαία αγορά, ενώ δεν αφορούν αυτές τις μικρομονάδες. Γι' αυτό πρέπει επιτέλους να καταλήξουμε κάπου με αυτή την μακρά ιστορία για τις μικρομονάδες, να κλείσει αυτή η ιστορία και η, αν περάσει με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, αυτό θα είναι πολύ θετικό για τις μικρομονάδες στην Ευρώπη. Επιτροπής για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές για το έργο που επιτέλεσαν τον Dirk Στέρ και τον κύριο Λένε. Πολύ σωστά το είπε ο κύριο Λένε, αυτό το σχέδιο της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιστοιχεί σε κάτι το οποίο είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 18 Δεκάτου του 2008 με ένα ψήφισμα και είχε πει ότι θέλει να κατεβάσει η Κομισιόν μια νομοθετική πρόταση ούτως ώστε τα κράτη-μέλη μπορούσαν να εξαιρέσουν αυτές τις μικρομονάδες από το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Επίσης να υπάρξει και κάποια ε, ε, ελάφρυνση όσον αφορά κάποιες διαδικασίε, διαδικασίες ώστε να μπορέσουμε να ωφελήσουμε αυτές τις εταιρείε και τέλος η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και αυτή συνέβαλε σε αυτή τη ε, διαδικασία της απλούστευτων λογαριασμών. Τώρα, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το νομοθέτημα, διότι θα πρέπει με ε, αυτόν τον τρόπο τα κράτη-μέλη να ομογενοποιήσουν αυτά τα οποία απαιτούνται από όλες ε, αυτές τις ε, μικρομονάδες και θα έχουμε μία μέθοδο αναφοράς ενιαία, είναι πάρα πολύ σημαντικό το μέτρο και αυτό θα ωφελήσει όσον αφορά τις σχετικές δαπάνες που κατέβαλαν αυτές οι μικρομονάδες. Έχουμε μια τάξη μεγέθους κάποιων δισεκατομμυρίων και θα φτάσουμε στα 6,3 δις ευρώ σαν οικονομίες όπως μου λένε οι υπηρεσίες πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα ποσά και αυτά βεβαίω βεβαίως δικαιολογούνται μια που θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στις οικονομικές δραστηριότητε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις και γι' αυτό και παρακαλώ να διεκπαιριωθεί ταχαίως αυτό το σχέδιο κειμένο και να εντάξουμε αυτό το νομοθέτημα στο, στο, πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τους λογαριασμούς ακριβώς όπως έχει συζητηθεί και από την Οικονομική Επιτροπή και έχουμε κάνει μια διαδρομή πολλών ετών μέχρι ότου μπορούμε να καταλήξουμε στην εφαρμογή αυτών των μέτρων. Θα λάβω υπόψη όλα αυτά τα οποία είπατε, αυτές τις παρατηρήσεις σας και ε, θέλω να σταθώ στα εξής τρία συγκεκριμένα σημεία. Πρώτα-πρώτα, με το σχέδιο κειμένου προσπαθούμε να δώσουμε το περιθώριο στα κρατημέλη για να μπορέσουν να διαλέξουν να κάνουν κάτι να μην το κάνουν δηλαδή μπορούν τους ισχύοντες κανόνες να τους διατηρήσουν ενισχύ και αν αλλάξουν το εθνικό τους δίκαιο τα κρατη δεύτερον αυτό το οποίο θέλουμε είναι το να ε, προστέψουμε την ομοθεσία να ε, προσφύγουμε στην επικουρικότητα γιατί δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κάποιους κανόνες κοινωτικού δικαίου και δεν επιβάλλεται. Και όσον αφορά τις μικρομονάδες έχουμε τώρα κάποιο πλέγμα και οτιδήποτε άλλο νομοθετήσουμε θα είναι περιττό. Επίσης δεν θέλουμε οποιαδήποτε διάταξη που διέπει τους λογαριασμούς και τα λογιστικά των μικρομονάδων να τις ε, καταργήσουμε ε, αποφάνθηκε από αυτό η νομική επιτροπή θα πρέπει βεβαίως να έχουν κάποια παραστατικά αυτές οι επιχειρήσεις ούτως ώστε να μπορούν να αποδείξουν το τι ε, ε, συναλλαγές έχουν κάνει και τα της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης παρακαλώ επιψηφίστε αυτό το κείμενο όλοι εμπλεκόμενοι τώρα περιμένουν την απόφαση και επομένως θα πρέπει να στείλουμε αυτό το μήνυμα από το Κοινοβούλιο να διεκπληρωθεί ο φάκελος είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει όλους αυτή η απλούστευση και φάνηκε από τη πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και επίση ελπίζουμε ότι οι μικρομονάδε άμεσα θα μπορούσαν να ωφεληθούν και να έχουν αυτή την εξοικονόμηση των παρών όπω θα γίνει με αυτό το νομοθέτημα. Οικονομικής και Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευτυχής που μπορούμε να παρουσιάσουμε εδώ στην Ολομέλεια την άποψη της Οικονομικής Επιτροπής. Ε, γιατί δεν ήταν και τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Ε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτή η ελάφρυνση για τις ε, μικρομονάδες. Νομίζω ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται διαφοροποίηση ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις και τις μικρές. Αλλά εδώ δεν νομίζω ότι επιτεύχθη ο στόχος. Εάν δεν υπάρξουν ετήσιοι λογαριασμοί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τι γίνεται, να έχουν πληροφορίες δηλαδή σχετικά με τους εμπορικούς τους εταίρους. Ε, δεν νομίζω ότι είναι καλό για τις ε, μικρομονάδες ε, οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις για αυτά τα θέματα. Σας ζητώ λοιπόν να ακολουθήσετε την άποψή μας και την πρότασή μας. Εμείς θέλουμε όχι μονάχα ε, ε, θετικά μέτρα, να σκεφτούμε λίγο και τα αρνητικά μέτρα. Θα πρέπει να δούμε και πώς εμπλέκονται οι οδηγίες ε, για, τα, για το δίκαιο των εταιριών και νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει διοικητική απλούστευση. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, γνωρίζουμε ότι οι μικρομονάδε είναι διαφορετικέ από τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και δεν μπορούμε να τι συγχαίουμε με τι μεγάλε επιχειρήσει. Αυτό θα είχε πολύ αρνητικέ επιπτώσεις, θα δημιουργούσε ένα αρνητικό περιβάλλον για τις μικρομονάδες και από πλευράς φορολογίας και από πλευράς γραφειοκρατίας και θα τους δημιουργούσε και μειωμένη ρευστότητα. Τα τελευταία χρόνια Αυτά τα μέτρα ήταν αποφασιστική σημασία για την ε, επιβίωση των μικρομονάδων. Ε, το 1 τρίτο ε, των μικρομονάδων δεν μπορούσαν να επιβιώσουν μέσα στην αγορά όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια. αν δούμε πόσο μεγάλο ποσοστό όλων των επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν αυτές οι μικρομονάδες, έχει σημασία να αρθούν όλοι οι φραγμοί, ιδίως ε, ε, να αντιμετωπιστεί το θέμα του διοικητικού φόρτου, της διοικητική επιβάρυνση για τις μικρομονάδες. Θέλουμε ε, όχι μόνο να απλουστεύσουμε τη διαδικασία για τις μικρομονάδες, ε, αλλά ε, πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε και το θέμα της κατάρτισης αιτήσεων λογαριασμών. Γιατί η κατάρτιση αιτήσεων λογαριασμών είναι μια απέτηση που αυξάνει το κόστος για τις μικρομονάδες και παράλληλα σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και το πώς θα απλουστεύσουμε τις ε, διαδικασίες της μικρομονάδες ε, που πρέπει να συντάξουν τους ή άλλως ε, λογιστικές καταστάσεις για φορολογικούς λόγους. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες απαιτήσεις για τις μικρές αυτές επιχειρήσεις. Πρέπει να δούμε και ποιο είναι το κόστος των νέων αυτών διατάξεων έχοντας κατά νου ότι αυτές οι επιχειρήσεις πολλές φορές είναι και μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Να μην επιβαρύνονται λοιπόν οι μικρομονάδες από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως ανέφερε και ο εισηγητής, αυτή η πρόταση οδηγίας αποτελεί συνέχεια ψηφοφορία στο Κοινοβουλίο, όπως επιθυμήσατε και εσείς κύριε Επίτροπε. Όμως ε, κριτικά βλέπει την πρόταση αυτή η ομάδα μου, γιατί κινδυνεύει να στραφεί κατά αυτών που θέλουμε να στηρίξουμε. Ε, θέλοντας ε, να ε, μειώσουμε το βάρος των επιχειρήσεων κινδυνεύουμε να τους αφαιρέσουμε στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για το δυναμισμό της δραστηριότητάς τους. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα κατόφλια και όσον αφορά το πώς ορίζουμε την μικρομονάδα μικρομεσαίες ε, ε, ε, πάνω, από 10 μέλη, 10 υπαλλήλους συγγνώμη, και πάνω από ένα εκατομμύριο τζίρο δεν μπορεί να μπαίνουν στις μικρομονάδες. Ενδεχομένως είναι ντόπιε και ενδεχομένως δεν είναι τόσο παρούσες σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Όμως πρέπει να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν για αυτές τις επιχειρήσεις να μην εφαρμόζονται οι λογιστικοί ε, κανονισμοί και να μην έχουν λογιστικές υποχρεώσεις ε, γιατί οπωσδήποτε έχει συναλλαγές με εμπορικούς εταίρους, ε, με τις ε, κοινωνικές και δημοσιονομικές αρχές, ε, με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστούν τους λογιστικούς κανόνες και εκεί ενδεχομένως να είναι πολύ πιο βαριοί οι κανόνες αυτοί. και τότε ενδεχομένως θα ε, εφαρμοστούν λογιστικές υποχρεώσεις πέρα και εκτός ε, των ε, ευρωπαϊκών πλαισίων και επομένως θα υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού και επομένως οι ευρωπαϊκές αυτές επιχειρήσεις θα υφίστανται διακριτική μεταχείριση. Τούτων λεχθέντων είναι σαφές ότι η απλούστευση των λογιστικών των μικρών επιχειρήσεων είναι ε, κάτι σημαντικό και υπάρχουν τρεις πρωτοβουλίες κατά αυτήν την έννοια. Η σημερινή πρόταση ε, το EFRS καθώς επίσης και η αναθεώρηση των ε, τέταρτης και έβδομης ε, οδηγίας που θα συζητηθεί σύντομα και άλλωστε αναμένουμε σύντομα και προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας τις είχαν υποσχεθεί για την αρχή του 2010, φαίνεται δεν θα τις έχουμε τόσο άμεσα. Εν πάση περιπτώσει εγώ δεν θα ήθελα, δεν θεωρώ μάλλον ότι ότι το ότι έχουν καθυστερήσει αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να μας οδηγήσει στο αντίθετο άκρο, ε, να επιταχύνουμε χωρίς λόγο τις διαδικασίες έτσι ώστε τελικά να μην επιτύχουμε τον επιδιωκόμενο στόχο. Πιστεύω κύριε Επίτροπε ότι θα ήταν καλύτερο και σαφέστερο για τις επιχειρήσεις να τους δοθεί μία ενιαία και συνολική ε, ε, απόφαση όσον αφορά την πραγματοποίηση ε, ακριβώς αυτής ε, της απλούστευσης που χρειάζονται οπωσδήποτε. Το παρόν πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστερεί να προτείνει αναθεώρηση των εν λόγω οδηγιών ε, και βεβαίως αυτό ε, αποτελεί πρόβλημα για μας. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να επιταχύνει τις συζητήσεις κυρίως όσον αφορά την εξαίρεση καθώς επίσης να κάνει και μελέτες αντικτύπου. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συναδέλφοι, ω και ηγήτρια συγγήτρια από την πλευρά των φιλελευθέρων, δεν καταλαβαίνω πώ θα μπορούσε να είναι κανεί κατά μια τέτοια διάταξη όταν μιλάμε για μικρομονάδε. Και τονίζω ότι είναι μικρομονάδε, όχι μικρομεσαίε. Δεν θα μπορούσαμε να διαφωνούμε από το να απαλλαγούν από τον φόρτο που επιβάλλει η κατάρτιση αιτήσεων λογαριασμών. Και από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από το κρατήδιο τη Βάδη Βιτεβέργη. Διακόπτεται η ομιλήτρια. Σα Σας είδα, αλλά σας είδα αργά, οπότε παρακαλώ να τελειώσει η κυρία και κατόπιν θα λάβετε το λόγο. Εάν δεχθεί ε, η ομιλήτρια που λάβει το λόγο την παρέμβασή σας. Και ευχαριστώ για τη συμβουλή σας. Προχωρήστε, συνεχίστε. Δεν μιλάμε για μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις από τη Βάδη με 100 εργαζομένους. Μιλάμε για ένα μικρό ανθοπολείο, για ένα μικρό φούρνο που προσπαθεί να επιβιώσει. Είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε τα τελευταία χρόνια, ακριβώς να απαλλάξουμε από αυτό τον επιπλέον γραφειοκρατικό ε, φόρτο της ε, μικρομονάδες. Είναι περί επιφόρτηση ε, γιατί θα πρέπει να καταφύγουν σε ειδικού που θα συντάξουν και θα ελέγξουν τους λογαριασμούς τους και θα πρέπει να τις διευκολύνουμε στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί πολύ καιρό προσπαθεί να πει στην Επιτροπή να καταλήξει σε μια πρόταση σαν αυτή την οποία έχουμε εδώ. Και από αυτές τις μικρομονάδες για τις οποίες συζητάμε μόνο το 7% έχουν διασυνοριακές δραστηριότητες. Επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα τήρηση της αρχής της επικουρικότητας και δεν υπάρχει επιβάρυνση της ενιαίας αγοράς από διαμεθοριακές δραστηριότητες των μικρομονάδων. Και επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για πολύ μικρές επιχειρήσεις και όχι για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν ακούμε ε, τα επιχειρήματα ότι μπορεί να ζητήσει μία πίστοση μικρομονάδα και να μην είναι δυνατόν να λάβει αυτή την πίστοση γιατί δεν θα υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα, ε, θα σας παραπέμψω στην ε, Βασιλεία 2. Και όσον αφορά το δεύτερο επιχείρημα για την προστασία των πιστωτών, θα να πω ότι ε, από την εμπειρία μου ως συμβολιογράφος ποτέ δεν είδα να αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα μια επιχείρηση που θέλει να συνεργαστεί με μια επιχείρηση που είναι τόσο μικρή όσο οι μικρομονάδες που συζητάμε. Και τρίτον, ε, όταν ε, μιλάμε για τις επιχειρήσεις αυτές ξέρουμε ότι μπορούν οι χώρες να κρατήσουν αυτές τις διατάξεις εφόσον μιλάμε για μια προαιρετική διάταξη. Ούτε ή άλλω θα πρέπει οι επιχειρήσει να τηρήσουν ε, τι απαραίτητε διατάξει όσον αφορά ε, την υποβολή ε, λογαριασμών για φορολογικού σκοπού. Παρακαλώ όλου λοιπόν να υπερψηφίσουν αυτή την πρόταση γιατί είναι αποτέλεσμα πολλών συμβιβασμών που έχουν γίνει για να καταλήξουμε στην Επιτροπή μας. Συνάδελφο, θέλω να σα υποβάλει μια ερώτηση. Αποδέχεστε την ερώτηση. Ναι. Ωραία. Έχετε μισό λεπτό. Κυρία, δέχεστε ότι θα πρέπει να καθυστερήσουμε αυτή την πρόταση για τη μελη των επιπτώσεων. Κάτι το οποίο είναι σαν να λέμε όχι. Έχετε 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε. Κατάλαβα την ερώτησή σας. Εάν η πρόταση αυτή απορριφθεί, τότε θα πρέπει να επανυποβληθεί και να την επανεπεξεργαστούμε και τότε ε, όντως ε, θα πρέπει να γίνει κάποια μελέτη αντικτύπου. Όπως είπα και προηγουμένως, βεβαίως ε, εμείς θέλουμε απλούστευση των λογιστικών των μικρομονάδων, ε, κυρίως ε, γιατί υπήρξε μια τέτοια συσσόρευση μέτρων και οδηγιών που σίγουρα πρέπει να αποσαφινιστεί η κατάσταση. Απλώς θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή δεν απλουστεύει τα πράγματα, αλλά αντιθέτως δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια στις επιχειρήσεις. Η κυρία Swinburne, για ένα λεπτό. Και νομίζουμε ότι επειδή έχει πάρα πολύ βελτίωση αυτή η πρόταση, εμείς ε, επιψηφίσαμε την πρόταση του κυρίου Στέρκη του εισηγητή, αλλά είπαμε ότι θέλουμε να καλέψει όλες τις μικρομονάδες της ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν για να τις βοηθήσει σε αυτά τα, τα έξοδα. Άρα χρειάζεται ε, να ξανααναθεωρήσουμε όλη αυτή την νομοθεσία και την τέταρτη και την πέμπτη οδηγίε για τι εταιρείε για να έχει νόημα αυτή η υπόθεση. Αυτή δε η πρόταση μας ε, προβληματίζει διότι από ό,τι φαίνεται είναι πολύ περιορισμένο το βελνικές τη πάντω, μέσα σε καιρού οικονομική κρίση οτιδήποτε βοηθάει οποιαδήποτε προσπάθεια έχει σημασία και στην Ουαλία, στην περιφέρειά μου νομίζω ότι οι ΜΜΕ κάπως θα ωφεληθούν και ε, βεβαίω δεν πρόκειται αυτό δεν είναι πανάκια γιατί του έχει χτυπήσει πολύ αυτή η ύφεση πάντω και αυτή η μικρή απαλλαγή ωφελεί της ε, επιχειρήσης, ιδίως αν συνεχίσει το έργο της ε, προστακή Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευτυχής κάθε φορά ε, που η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπονεί κάποιο σωστό κανόνα, αλλά ε, ξέρετε ε, τελικά δημιουργείται ένα ιδιαίτερα σφιχτό πλέγμα κανόνων που δυσκολεύει τη ζωή των ε, ανθρώπων. Είναι γεγονός ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί ε, ε, είναι απαραίτητοι έτσι ώστε να υπάρξει η απαραίτητη διαφάνεια στον χρηματοπιστωτικό τομέα και γενικότερα στους εμπορικούς λογαριασμούς. Βεβαίως για τις μικρομονάδες τα πράγματα πρέπει να είναι λίγο διαφορετικά. Όμως εάν ε, από τη μία πλευρά απλουστεύουμε και από την άλλη πλευρά ε, ε, επιβάλλουμε νέους κανόνες, τότε αναρωτιόμαστε μήπως τελικά το βάρος είναι μεγαλύτερο. Θέλουμε οι δηλώσεις να ελέγχονται 100% να έχουν διαφάνεια πλήρη έτσι ώστε και οι μικρομονάδες να ξέρουν τι τους περιμένει. Νομίζω ότι εδώ ε, αναφερόμαστε σε μέτρα τα οποία θα είναι ικανοποιητικά για πολλές μικρομονάδες και επομένως ε, θα είναι πολύ καλό για την οικονομία γενικά. Ε, Έχουμε φτάσει στο 20% στον αφορά την ενεργεία στους νέους στην Ηνωμένο Βασίλειο και στην Γαλλία η ενεργεία στους νέους είναι 24% από την άλλη μεριά. Μιλάμε για 25% στην Ιταλία και το τρομερό 39% έχει χτυπήσει στην Ισπανία. Οι δε μεγάλες εταιρείε τελευταία γιατί απολύουν συνέχεια εργαζόμενους και θα συνεχίσουν αυτή την πορεία τους. Επομένως για τους ανέργους η ελπίδα είναι οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικρομονάδες. Όμως οι οδηγίες της ΕΕ δυσκολεύουν την ε, εύρυθμη λειτουργία αυτών των εταιριών και επίσης από τους κανονισμούς της ε, ΕΟΚ ασφικτιούν αυτές οι ίδιες εταιρείε. Ε, οπότε θα πρέπει να βγει κάτι λογικό ε, από την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. οπότε από αυτούς τους λογαριασμού εταιριών να απαλλαγούν αυτές τις εταιρείε. 1,7 εκατομμύρια έχουμε μικρές μονάδες στη χώρα μας οπότε εάν μπορέσουν έναν, έναν μόνο να απασχολήσουν παραπάνω τότε ε, το πρόβλημα της ενεργείας στη χώρα μας θα επιληθεί. Όλοι λάβαμε αυτό το κείμενο του κ. Στέρξη και της παρέας του και ποντάρουν στο ότι εάν απαλλάξουν αυτές τις μικρές επιχειρήσεις αυτό θα είναι κάτι το οποίο αντιβαίνει στην ιδέα της ενιαίας αγοράς. Είναι γελίος αυτός ο ισχυρισμός που μόνο ένας φιλελεύθερος Βέλγος θα μπορούσε να διανοηθεί. Και εδώ στο κοινοβούλιο βέβαια, όποιο πει τίποτα κακό για του Βέλγους, τρώει πρόστιμο. Αλλά πριν από 96 χρόνια, εμεί δώσαμε μάχη. Μάχη και πολεμήσαμε για να προστατεύσουμε την αναδευτική ακυρότητα του Βελγίου. Οπότε α λογικευτεί αντίστοιχα ο κύριο Στέρξ και α μην χτυπάει την οικονομία τη δική μου χώρα. Ε, για Uh, Εάν πραγματικά θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο, κύριε Στέρξ, εντάξει. Αλλά περιμένετε λίγο. The Earl of Dart, uh, uh mm, mm, ο Earl of Dart σας έχει υποβάλει μια ερώτηση. Ναι, ε, φαντάζομαι ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής και ευγνώμων για ό,τι έκανε η Βρετανία πριν μερικά χρόνια για μας. Αλλά μια ερώτηση. Φέτος προγραμματίζει αναθεώρηση δύο οδηγιών ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν λοιπόν αναθεωρηθούν ε, οι δύο οδηγίες, πιστεύετε ότι θα αντιταχθούν στο σκοπό που έχουμε για απλούστευση των κανονισμών. Απάντηση οι μικρές επιχειρήσεις θέλουν, χρειάζονται απλούστευση των λογιστικών τους τώρα. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Λένε για την εξαίρετη έκθεση που μας υπέβαλε. Τον ευχαριστώ ε, για τον, ε, για την ικανότητα διαλόγου ε, και την ε, πεποίθηση που έχει όσον αφορά τον αγώνα για τη διευκόλυνση των μικρών επιχειρήσεων. Γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα. Και η πρόταση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρίως σε όρους κρίσης Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να εξακολουθήσουν να υφίστανται ανώφελες υποχρεώσεις. Θα πρέπει να διατηρηθούν μονάχα οι υποχρεώσεις αυτές οι οποίες αφορούν τη διαφάνεια ε, και που ε, αφορούν ε, τελικά την επιβίωση και την σωστή παρουσία των μικρομονάδων, των μικρών επιχειρήσεων. Δεν είναι δυνατόν να βάλουμε στο ίδιο καλάθι διαφορετικές επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν να απευθυνόμαστε με τον ίδιο τρόπο και να απαιτούμε τα ίδια πράγματα από τελείω διαφορετικέ μεταξύ του ε, επιχειρήσει. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να βοηθήσουμε τι μικρομονάδε αυτέ, ε, οι οποίε μπορούν, εάν βοηθηθούν, να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξη. Δυστυχώς στην Ευρώπη, στις χώρες μας βλέπουμε κάθε μέρα να κλείνουν τέτοιες μικρές επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Οι ε, ε, ε, προτάσεις που γίνονται εδώ είναι αντίστοιχες με κάποιες προτάσεις που είχαμε στο Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ τουλάχιστον και από τους συναδέλφους τους Πορτογάλους να προσπαθήσουν να ξεπεραστούν ε, τα προβλήματα τα οποία έχουν μπλοκάρει ε, το θέμα στο Συμβούλιο και μάλιστα η χώρα μου, η Πορτογαλία, μπλοκάρει ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ κύριε ο στόχος της ε, μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης για τις μικρομονάδες ε, σαφώς είναι ο στόχος που μας βρίσκει σύμφωνος. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τις μικρομονάδες βάζοντάς σε στην ίδια κατηγορία με τις μεγάλες επιχειρήσεις για την κατάρτιση ετησίων λογαριασμών. Μπορεί όμως αυτό να επιτευχθεί με την πρόταση της Επιτροπής και σύμφωνα με την ε, πρόταση του κ. Λένε. Η Χωνσός Καστέξ ήδη ανέφερε το θέμα των μικρών επιχειρήσεων ή μικρομονάδες. Είναι ε, πολλές φορές όχι τόσο μικρές. Πρόκειται για εταιρείε περιορισμένες ευθύνης πολλές φορές στην Αυστρία και μπορεί το 90% όλων των επιχειρήσεων που έχουν κάτω από 10 ε, υπαλλήλους να εντάσσονται σε αυτή την ε, κατηγορία. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής ετήσιων λογαριασμών. Ε, αντί να απαλλαγούν από την τέταρτη οδηγία οι μικρομονάδες, θα έπρεπε να συνταχθεί ε, νέα οδηγία, να συνταχθούν νέες διατάξεις ε, για να εξαιρούνται από τις περιττές υποχρεώσεις οι μικρομονάδες. Ευχαριστώ. Ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η οικονομική κρίση δείχνει σαφώ ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να συνεχίσει να συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη σε άλλα μέρη του κόσμου και με την οικονομική ανάπτυξη τη Ασία, παραδείγματο χάρη. Η δομή της ε, δικής μας κοινωνίας ε, διαφέρει κατά πολύ. Πόσο ε, πώς μπορούμε να συγκριθούμε με τους εργαζόμενους στις χώρες της Ανατολικής Ασίας ε, στην ε, Κίνα. Στις χώρες μας υποχρεώνονται οι εργαζόμενοι να υποβάλουν δηλώσεις σε τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις, σε τέσσερις διαφορετικές υπηρεσίες, στην οικονομική φορολογική υπηρεσία, στη στατιστική υπηρεσία, σε υπηρεσίες για κοινωνική και για κοινωνική ασφάλιση και για άλλα κοινωνικά δικαιώματα. Ε, και οι επιβαρύνσεις, οι διοικητικές αυτές ε, επιβαρύνσεις από κρατικούς φορείς ε, είναι ε, πολύ μεγάλη επιβάρυνση για τις μικρομονάδες από τις οποίες απαιτούν πάρα πολύ χρόνο και προσπάθεια. Θα μπορούσαμε είτε να άρουμε αυτές τις περιττές διατάξεις για να γίνουν πιο αποτελεσματικές οι διατάξεις για το διοικητικό φόρτο ε, είτε να καταστρέψουμε το μέλλον αυτών των επιχειρήσεων και νομίζω ότι θα έπρεπε να επιλέξουμε την πρώτη λύση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ήμουν και εγώ στην ε, ομάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολλοί από εμά έχουμε συνεργαστεί για το Small Business Act, ε, αυτή την πρωτοβουλία για τις ε, μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και ξέρουμε ότι η πρωτοβουλία έχει σαν προσταγή το ότι πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία ακούσαμε φαίνονται πάρα πολύ ελκυστικά. Αν ήταν τόσο ελκυστικά, γιατί να μην χειροκροτούν όλες οι πλευρές αυτή την πρωτοβουλία, γιατί υπάρχουν τόσο διαφορετικά παραδείγματα σε αυτόν τον τομέα και γιατί υπάρχουν τόσο πολλές και διαφορετικές φωνές και δεν συμφωνούν και δεν χειροκροτούν όλοι. Είναι συμβατό με την Βασιλεία 2 από τη μια πλευρά προσπαθούμε να έχουμε κοινέ διατάξεις για τη σύνταξη ετησίων λογαριασμών και από την άλλη πλευρά προσπαθούμε να καταργήσουμε αυτή την υποχρέωση τήρησης ευρωπαϊκών ετησίων λογαριασμών. Θέλουμε να έχουμε ευρωπαϊκές λύσεις, όχι εθνικές λύσεις. Δεν θέλουμε να έχουμε κατακαιρματισμό ε, του δικαίου και δεν θέλουμε να έχουμε διαφορετικές διατάξεις η απελευθέρωση αυτών των μικρομονάδων από τη σύνταξη ετησίων λογαριασμών δεν θα ήταν τελικά ε, ε, απαλλαγή από επιπλέον φόρτο, γιατί τα ίδια δεδομένα θα έπρεπε να τα δίδουν σε πολλές χώρες για διαφορετικούς σκοπούς. Αλλά θα ήταν πιο δύσκολη η επιτήρηση, θα ήταν πιο δύσκολο να γίνει ο έλεγχος. είναι διατάξεις που πρέπει να τηρούνται και από τις μικρές επιχειρήσεις για να μην χάνεται η διαφάνεια. Για να μπορέσουν να μεγαλώσουν αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρήσουν κάποιες διατάξεις και θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής στα κράτη-μέλη, πράγμα το οποίο αποδυναμώνει την ενιαία αγορά. Εγώ είμαι υπέρ του να επανεξεταστούν οι οδηγίε πλαίσιο, η τέταρτη και η έβδομη οδηγία, ούτω ώστε να καταλήξουμε σε ενιαίε διατάξει που θα οδηγήσουν στην ελάφρυνση των μικρών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι θέλουμε να μειώσουμε το διοικητικό βάρος και πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ε, πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, οι οποίες είναι αυτές που υποφέρουν περισσότερο. Όμως δεν πρέπει να τα πετάξουμε όλα καλά και άσχημα μαζί Δηλαδή, ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες ε, αρχές. Ε, υπάρχουν κάποιες ε, επιχειρήσεις οι οποίες αφορούνται περισσότερο από το θέμα των διακινητικών ανταλλαγών. Υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις οι οποίες στις διασυνοριακές τους ανταλλαγές αντιμετωπίζουν προβλήματα. Υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κεντρική έδρα και θυγατρικές. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Ε, όσον αφορά τώρα τη διαφάνεια βεβαίως όλοι τη θέλουμε και οι ίδιες οι επιχειρήσεις ε, και οι συνδικαλιστέ. Ε, οι ίδιες οι επιχειρήσεις θέλουν να ξέρουν πώς λειτουργούν και με το, για, να ξέρουν ακριβώς πώς λειτουργούν και για να ξέρουν πώς λειτουργούν και οι ενδεχόμενοι εμπορικοί του εταίροι χρειάζονται καθαροί λογαριασμοί σε πολλές ε, χώρες της Ευρώπης ε, οι μικρές ε, επιχειρήσεις έχουν φόβους όσον αφορά την κατάσταση και τις, τα μελλοντικά προβλήματα τα οποία ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Εκτιμώ απεριόριστα την εργασία του συναδέλφου Λένε, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ την έκθεση αυτή. Συμφωνώ όμως με τις προτάσεις Στέρξα, δηλαδή να αξιολογήσουμε τα πάντα ε, και να προχωρήσουμε μετά σε μια συνολική αναθεώρηση ε, ε, των οδηγιών για το δίκαιο των εταιριών. Είχε αναγγελθεί για φέτος αυτή η αναθεώρηση και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να αργήσει. Okay. <laughs> Ε, δεν είχα ακούσει το όνομά μου, ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Νομίζω ότι ε, ήδη ελέγχθησαν τα πιο σημαντικά σχετικά με αυτή την οδηγία. Νομίζω κανείς σε αυτήν την αίθουσα δεν μπορεί να ε, διαφωνεί με την μείωση των διατάξεων που επιβαρύνουν τις μικρομονάδες πρέπει να δούμε μέχρι που θέλουμε να φτάσουμε γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε διατάξεις για την κατάρτιση ε, λογαριασμών και θα πρέπει και οι μικρομονάδες να τηρούν λογαριασμούς για να μπορούν να αποδείξουν την οικονομική τους θέση και σύμφωνα με το Βασιλεία 2 υπάρχουν διατάξεις, επομένω δεν προτείνεται τίποτα ε, νέο σε σχέση με διατάξεις ε, που υπάρχουν και τηρούνται και σε άλλες ε, χώρες. θα πρέπει να είναι δυνατόν μέσα σε ένα χώρο ανταγωνισμού όπως ε, η Ευρώπη να υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και νομίζω ότι όλοι αυτό θα θέλαμε όχι μόνο για τις μικρομονάδες αλλά και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν τέτοιες ενιαίες διατάξεις. Ε, σίγουρα χρειάζεται υποβολή των δεδομένων, υπομορφή λογαριασμών, υπομορφή παροχής άλλων δεδομένων. Και οι μικρομονάδες δεν μπορούν να υποβάλουν τα ίδια στοιχεία που υποβάλλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα στο πλαίσιο της τέταρτης και της έβδομης οδηγίας, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα απαλλάσει πραγματικά από την ε, επιπλέον ε, επιβάρυνση της μικρομονάδα. Εάν θέλαμε να ξεκινήσουμε μια εταιρεία, μάλλον οποιοδήποτε μα το έκανε θα έφτιαχνε μια μικρομονάδα Χρειαζόμαστε νέες επιχειρήσεις. Γιατί σοβεί μια κρίση και μας έχει χτυπήσει και η ανεργία και για να την αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να φτιάξουμε όσο γίνεται περισσότερες μικρομονάδες. Μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή μικρομονάδες και επομένως θα πρέπει ό,τι πέρα από το χέρι μας το κάνουμε, τόσο ώστε να δώσουμε κίνητρα για να δημιουργηθούν τέτοιες επιχειρήσεις. Αυτό κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της. Προσπαθεί να τις ε, απαλλάξει από αυτούς τους αιτήσους λογαριασμούς. Και για τρεις λόγους θα πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα-πρώτα, γιατί όπως προείπα στην πράξη οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις ξεκινούν την εταιρική ζωή τους ως μικρομονάδες. Επομένως, με την ε, σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δούμε αν τα πράγματα θα πάνε καλύτερα γιατί δεύτερον το, οι δαπάνες για τους ετήσιους λογαριασμούς δεν είναι δυνατόν να ε, συγκριθούν με τα κέρδη. Τα κέρδη και για την εταιρεία αλλά και για το κράτος γιατί αν κανείς τη χρειάζεται πίσω σε μια τράπεζα τότε θα πρέπει κανείς να έχει την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση και θέση της εταιρεία και όχι κάτι το οποίο ε, συντάχθηκε πριν από ένα χρόνο και επομένω. Ε, λέμε τώρα για μείωση του, των διοικητικών δαπανών κατά 25% αυτό θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για όλους αυτούς τους λόγους σας λέω, ας σταματήσει μια τέτοια συζήτηση για η στήριξη των επιχειρήσεων. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσουμε τα λόγια και να πάμε στα έργα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει όλο ένα και αυξανόμενη θέση και πιο σημαντική θέση στο ευρωπαϊκό πανόραμα, αλλά παρόλα αυτά ε, δεν έχουμε δει μέτρα τα οποία να τις ευνοούν. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάποιες ε, προτάσεις τύπου small business first έτσι ώστε να να βελτιωθεί η παρουσία αυτών των μικρών επιχειρήσεων στον επιχειρηματικό κόσμο η απλούστευση των λογαριασμών τους, ε, η διευκόλυνση της εισδοχής τους ε, στον εμπορικό κόσμο ε, είναι οπωσδήποτε πολύ θετικά στοιχεία. Ο κύριος Λένε οδηγείται ε, στο συμπέρασμα ότι θα ευνοηθούν αυτές οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από τις διοικητικές απαλλαγές ε, που προτείνονται. Βεβαίως εμείς θα θέλαμε να δούμε ε, και μεγαλύτερη εναρμόνιση στον, ε, στο, στον νομικό ε, τομέα. Βεβαίως θέλουμε επίσης να δούμε την αναθεώρηση των οδηγιών που αφορούν τις ε, εταιρείε. Και βεβαίως εγώ ερχόμενη από μια χώρα η οποία έχει μνημειώδη γραφειοκρατία πραγματικά θα συμφωνήσω πλήρως με την απλούστευση και την μείωση των επιπλέον επιβαρύνσεων πλαίσιο για τις μικρές επιχειρήσεις. του Έχω έξι ομιλητές και αυτοί οι έξι θα μιλήσουν ε, και μόνον. Η κυρία Χολμάιερ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μου κάνει εντύπωση η συζήτηση από πλευρά των συναδέλφων ε, που εδώ αφενό με μιλούν υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη απλούστευσης. Ε, από την άλλη πλευρά δεν κάνουν το πρώτο βήμα για τις μικρομονάδες για τις οποίες μιλάμε σήμερα. Γιατί σήμερα μιλάμε για τις μικρομονάδες και όχι για μεγάλες ε, επιχειρήσεις. Έχω μιλήσει με πολλές μικρομονάδες και από τις μικρομονάδες αυτές έχω ακούσει ότι ελπίζουν ακριβώς την ψήφιση αυτών των διατάξεων για την ελάφρυνση ε, της, ε, των επιβαρύνσεων για αυτές τις μικρομονάδες. Δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά την διαφάνεια, διότι υπάρχουν οι διατάξεις, όπως πολύ σωστά είπε και ο Επίτροπος, θα παραμείνουν οι διατάξεις που θα εξασφαλίζουν περαιτέρω τη διαφάνεια. Εξάλλου, αυτές οι διατάξεις για τις μικρομονάδες δεν έχουν επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή αγορά, γιατί δεν ασκούν διευρωπαϊκό εμπόριο αυτές οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό παρακαλώ τους συναδέλφους να ψηφίσουν υπέρ της έκθεσης του κ. Λένε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκοζές για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ με τα περισσότερα από τα επιχειρήματα που ακούσαμε, την Μαρία Τάισεν, τον κύριο Καράσεν, την κυρία Καστέξ και αναρωτιέμαι, θα πρέπει μετά από αυτή τη συμβαστική ε, τροποποίηση να αφήσουμε τις εθνικές επιλογές και έτσι να μπλοκάρουμε αυτή την ε, οδηγία που είναι ένα μήνυμα θετικό και απλούστευσης προς τις μικρές επιχειρήσεις. Επίτροπε, εγώ σας προτείνω το εξής. Πρώτα, πρώτα ε, θα πρέπει να επιψηφίσουμε την πρόταση Λένα και θα πρέπει και εσείς ο ίδιος να λάβετε υπόψη σοβαρά αυτό το οποίο είπαμε για τις τροποποίησεις των άλλων δικαιών ώστε ταχύως να μπορέσουν να προχωρήσουμε προς μια εναρμόνιση κυρίως όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν τους λογαριασμούς και τα λογιστικά των εταιριών. Κέλλη, όπως και άλλοι συνάδελφοι, στις 4 η ώρα ξημερώματα σηκώθηκε για να έρθω εδώ, αλλά με μεγάλη μου χαρά. Ακόμα εδώ ξενυχτάω γιατί είναι γεμάτες ελπίδα αυτά, τα οποία συζητούμε. 7,6 δις θα είναι η εξοικονόμηση από αυτή την απαλλαγή και είναι πολύ σημαντικό. Οπότε αυτό απαντά σε κάποιες επικρίσεις. Ότι δηλαδή είναι πάρα πολύ γραφειοτική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως κάνουμε διορθωτικές κινήσεις στα στραβά που υπάρχουν γιατί οι τράπεζες από την άλλη μεριά ούτε καμία ενοχή φαίνεται νιώθουν ούτε κάνουν τίποτε. Θα πρέπει επομένω να δούμε τι θα κάνουμε για να φτάσουμε τόσο 85% και αυτό να το κάνουμε το συντομότερο. για ένα λεπτό. Πολύ, κύριε Πρόεδρε. Διανύουμε περίοδο οικονομικής κρίσης και είναι δεδομένο ότι η απαλλαγή των μικρομονάδων από την εκ του υποχρέωσή τους να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν ετήσιους λογαριασμούς είναι ένα ευπρόσδεκτο μέτρο στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και βεβαίως στο σημείο αυτό συμφωνώ με τον εισηγητή. Και είναι γεγονός πως μια τέτοια ενέργεια μειώνει το λειτουργικό κόστος των εταιριών, αυξάνει την κερδοφορία τους και ενδεχομένως συμβάλλει θετικά στη διατήρηση θέσεων εργασία. Ωστόσο, και νομίζω εδώ είναι η ανησυχία ε, αρκετών συναδέλφων, ε, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο και τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να δώσουμε άμεσα και γρήγορα ανάσα στον ευαίσθητο αυτό οικονομικό τομέα. στόχος θα πρέπει να είναι η ανακούφιση και όχι και σε αυτό θέλω να δώσω έμφαση η παροχή άλοθη προς αυτές τις επιχειρήσεις για την παραποίηση ή απόκρυψη των πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καλή ε, περαιτέρω πορεία τους. επομένως λοιπόν καταρχήν νομίζω πρέπει να χαιρετήσουμε και να υποστηρίξουμε με θέρμη την πρόταση της επιτροπής και βεβαίως να είμαστε προσεκτικοί στις ρυθμίσεις που λαμβάνουμε και στο μέλλον για να μην αλλοιώνονται οι πραγματικές μας προθέσεις η στήριξη δηλαδή αυτών των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Μπαλσίτης, για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σίγουρο ότι πρέπει να είναι σίγουρο ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τις μικρομονάδες και ένα από τα καλύτερα μέσα που διθέτουμε είναι η μείωση της φορολογίας για τις μικρομονάδες και η διευκόλυνση αυτών των επιχειρήσεων στις ορισμένες υποχρεώσεις τους. Ακούστηκαν κάποιες ιδέες σήμερα. Όταν κάποιος θέλει να πάρει μια πίστοση από τράπεζα, θα πρέπει να υποβάλει κάποιες πληροφορίες στην τράπεζα. Ε, κάποιες είναι αυτονόητες, κάποιες άλλες είναι συμπληρωματικές. Αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες αντιστοιχούν σε μια επιπλέον επιβάρυνση. Η απαλλαγή των μικρομονάδων από την υποχρέωση αιτήσεων λογαριασμών, κατά τη γνώμη μου, είναι θετικό και θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις. Είναι εδώ η κυρία Τάιν. Ωραία. Λοιπόν, εξ ονόματος της Επιτροπής, ο κύριος Μπαρνιέ, παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρά το προκεχωρημένο της ώρας, ε, αναφερόμαστε εδώ σε ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Άκουσα όλες τις απόψεις όλων όσων εκφράστηκαν εδώ. Και όλοι οι βουλευτές αναφέρθηκαν στην ανάγκη μείωσης του διοικητικού άχθους των μικρομονάδων, των μικροεπιχειρήσεων. Περίπου 5 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην Ευρώπη ενδεχομένως θα αφορά ε, αυτό το κείμενο από ό,τι μου είπαν ε, οι συνεργάτες μου. Υπάρχουν βεβαίως κάποιες ε, αποκλήσεις όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και ε, όσον αφορά ή όσον αφορά ε, τον τρόπο εφαρμογής. Γνωρίζετε ποια είναι η άποψή μου. Έχω εκφραστεί επανειλημμένα και όταν μάλιστα είχατε την καλοσύνη να οργανώσετε την ακρόασή μου αναφέρθηκα και σε αυτό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει οι ε, μικρές επιχειρήσεις να βρουν πρώτα τη θέση τους μέσα στα πλαίσια αυτής της μεγάλης οικονομικής ενιαίας αγοράς. Χρειάζεται μεγάλη αποφασιστικότητα. Βεβαίως μπορεί περαιτέρω να βελτιωθεί το κείμενο αυτό. Όμως, πιστεύω, όπως είπε και ο πρόεδρος λένε, ότι οφείλουμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα ε, προς τους ε, ενδιαφερόμενους. Ε, με μεγάλη ευχαρίστηση άκουσα ένα σπάνιο σχόλιο θετικό προς την Κομισιόν η οποία αναγνωρίζεται ότι για μία φορά τουλάχιστον ότι κάτι καλό προσπαθεί να κάνει. Όμως πρέπει να σας πω ότι πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει συγκεκριμένα απτά λογικά ε, και ωφέλιμα πράγματα και ευελπιστώ ότι και στο μέλλον θα έχω τη δυνατότητα να σας το αποδείξω έτσι ώστε να σας πείσω ότι σε όλα τα μέτωπα η Κομισιόν προσπαθεί ε, να είναι ε, σωστή και χρήσιμη. Και βεβαίως ε, πάντα με τη στήριξη και συχνότατα μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η πρόταση αυτή είναι συγκεκριμένη, είναι βαθμιαία είναι λογική και επομένως με τρόπο πολύ λογικό απλουστεύει ε, το διοικητικό άχθος των μικρών επιχειρήσεων. Δεν, δεν έρεται με κανένα τρόπο η υποχρέωση υποβολής λογιστικών καταστάσεων, λογαριασμών και επομένως ε, ε, θα ήθελα με τον τρόπο αυτό να απαντήσω και στις ανησυχίες του κυρίου Στέρξε. Βάσει της προτάσεως, αυτών, της προτάσεως αυτής ε, θα, βελτιωθεί, θα βελτιωθούν οι κανόνες, οι λογιστικοί σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο δηλαδή στο επίπεδο που εργάζονται ε, αυτές οι επιχειρήσεις, σε το τοπικό επίπεδο. Βεβαίως και το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει η εφαρμογή να γίνει όσο γίνεται πιο ε, γρήγορα. Νομίζω ότι το οφείλουμε αυτό στις μικρές επιχειρήσεις. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την κυρία Κάστεξ να αναφέρεται σε αυτόν τον επόμενο ορίζοντα ε, στις μελλοντικές χρονικές στιγμές της ε, των αναθεωρήσεων των ε, οδηγιών. Οι προθεσμίες ε, επί των οποίων εργαζόμαστε, ενδεχομένως να μην είναι το τέλος του 2010 που αναφέρατε εσείς, να είναι το 2011, μας οδηγούν στο συμπέρασμα και να πω εδώ ότι εν παρόδο ότι άκουσα ε, την σαφή παρένεση του κυρίου Γκοζές. Ε, ναι, ε, βεβαίως εμείς θα κινηθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι πραγματικά δεν υπάρχει καμία συμβατότητα ανάμεσα στο να εφαρμοστεί αμέσως η πρόταση για τις μικρομονάδες αμέσως τώρα και μετά αργότερα να προχωρήσουμε με άλλες βελτιώσεις στα πλαίσια της συνολικής αναθεώρησης ε, της οδηγίας για τους λογαριασμούς. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Απλώς το δεύτερο σκέλος θα πάρει λίγο χρόνο ακόμα. Και πιστεύω ειλικρινά ότι λαμβάνοντα υπόψη την παρούσα κατάσταση πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα πολύ συγκεκριμένα πράγματα που είπαν και ε, ο κύριος Ντεγιόγκ και ο κύριος Φεγιό και άλλοι ε, βουλευτές που αναφέρθηκαν στην κρίση την οποία διανύει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Βάσει των υπολογισμών μας καταδεικνύεται ότι βάσει αυτής της τροποποίησης, αν εφαρμοστεί αμέσως, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να βοηθήσουμε άμεσα την ανάκαμψη της οικονομίας. Βάσει και των προτάσεων ε, Μπαρόζο. Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο θα κάνει πιο αποτελεσματική την αγορά και βάσει αυτών των μέτρων μπορούμε μόνοι μας ε, να έχουμε αύξηση της ε, ε, παραγωγικότητας, να έχουμε ανάπτυξη από 0,5 έως 1,5%. Και γιατί να ε, προσπαθήσουμε απ' έξω να βρούμε αυτήν την ανάπτυξη τη στιγμή που η ανάπτυξη υπάρχει σε αυτές τις 5 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Αυτή είναι η φιλοσοφία λοιπόν της πρότασής μας. Άκουσα τον κύριο Κάρας, την κυρία Ράνερ ε, και άλλους ε, να αναφέρονται στα, στα ελάχιστα στάνταρ, στις ελάχιστες απαιτήσει και άλλωστε η έκθεση του κυρίου Λένε δεν κλείνει την πόρτα σε τέτοιου είδους ε, ελάχιστες απαιτήσει. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κατά αυτή την έννοια και με το Συμβούλιο αλλά σας παρακαλώ ασχοληθείτε με την έκθεση αυτή, δέστε ότι η έκθεση αυτή, δέστε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ε, κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρώτο θετικό βήμα ε, υπέρ όλων αυτών των μικρομονάδων που παλεύουν να αντιπαρέλθουν ε, τις δυσκολίες οι οποίες είναι ακόμα περισσότερες τώρα σε αυτήν την ε, κατάσταση κρίσης. και δεσμεύομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου να δουλέψουμε όσο γίνεται πιο ε, γρήγορα μαζί με το Συμβούλιο έτσι ώστε να δώσουμε στις μικρές επιχειρήσεις τη θέση τους σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τον κύριο Επίτροπο για την συνέχιση. Έχω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Πρώτον για την αξιολόγηση επιπτώσεων. Η Επιτροπή έχει κάνει μια εκτενέστατη αξιολόγηση επιπτώσεων και στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων μετά την παρουσίαση της έκθεσης ΣΤΕΡΚ από την Επιτροπή Νομικών, Οικονομικών Υποθέσεων ε, εξετάσαμε τα θέματα των ε, επιπτώσεων. Μέχρι τώρα δεν λάβαμε απάντηση ε, για το θέμα αυτό. Ε, δεύτερον, μιλάμε για μια συμβαστική λύση που αποτελεί τις ελάχιστες διατάξεις. Δεν μιλάμε για μείωση των υποχρεώσεων για τα στοιχεία τα οποία πραγματικά είναι απαραίτητο να υποβάλουν οι επιχειρήσεις. Ε, τρίτον, όποιος χρειάζεται ένα τέτοιο ισολογισμό για την λήψη τραπεζικής πίστοσης μπορεί να καταρτήσει ένα τέτοιο ισολογισμό. Αλλά επιχειρήσεις που δεν χρειάζονται ένα τέτοιο ισολογισμό, γιατί να τις επιβαρύνουμε με μια επιπλέον διάταξη. Τέταρτον, ε, οι διατάξει ε, κατάρτιση δεδομένων για φορολογικού ε, σκοπού παραμένουν ενισχύει απλώς δεν επιβαρύνουν περαιτέρω τις επιχειρήσει επόμενο σημείο. Δεν είναι μικρό έργο η αναθεώρηση της τέταρτης και της έβδομης οδηγίας. Είναι ένα γιγαντιαίο έργο. Είναι ένας τομέας πάρα πολύ ε, πολύπλοκος ε, και ε, τολμώ να προβλέψω ότι αν τώρα λάβουμε μια τέτοια απόφαση θα υπάρχει ο κίνδυνος μιας μεγάλης αναθεώρησης της τέταρτης και έβδομης οδηγίας αλλά μέχρι τότε θα έχουν καταποντιστεί οι μικρομονάδες γιατί δεν μπορούν να παίξουν ένα ρόλο μέσα σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Είναι σημαντικό η απόφαση αυτή λοιπόν για τις μικρομονάδες να ληφθεί τώρα και να μην περιμένουμε για αργότερα που ακόμη δεν ξέρουμε πότε θα σημαίνει και προς τα που θα κινηθούμε. Επόμενο σημείο. Νομίζω ότι όλοι είναι υπέρ αυτή τη ε, διάταξη εκτό από κάποιε μεγάλε επιχειρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Στον εισηγητή η συζήτηση έληξε ψηφοφορία Τετάρτη στι 12 το μεσημέρι. Και περνάμε τώρα στην τελευταία συζήτηση της διάταξης, ε, που είναι η σύντομη παρουσίαση της έκθεσης της κυρίας Ίντβελ σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού του 2008. Ε, έχω την ε, ευχαρίστηση να σας ανακοινώσω ότι αυτή η συζήτηση περιέχει μόνο